Παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας, κυρίες και κύριοι. Ich Υπενθυμίζω ότι δυνάμη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού υπό την Προεδρία του αποχωρούντος Προέδρου δεν γίνονται ομιλίες οι οποίες να μην έχουν σχέση με την εκλογή νέου Προέδρου ή το περιεχόμενο της εντολής του. Δηλαδή ομιλίες, παρεμβάσεις δεν θα γίνουν δεκτές πέραν αυτών που αφορούν την συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Έχουμε λοιπόν για σήμερα στην εμερήσια διάταξη την έκκληση, την εκλογή συγγνώμη του ητής Προέδρου δυνάμει του κανονισμού. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου κατατίθενται δυνάμει του άρθρου 15